Ναι, φυσικά ε, δεν ήταν σωστό αυτό που υπόθηκε. Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω ε, αντιπροσωπεία του Κυρκιστάν ε, που βρίσκονται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κυρκιστάν. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ευχόμαστε να έχετε μια επικοδομητική συζήτηση σήμερα. Έχω λάβει την θέση του Συμβουλίου ε, στην πρώτη ανάγνωση σχετικά με το dumping και τις ε, ενισχύσεις από πλευράς ε, μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.